Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 5η για το θέμα αυτό. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο 9 με 1 και 3 με 7. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί στο ε, έγγραφο συνεδρίας και στο ίντερνετ. Λύεται η συνεδρία.